Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σε ένα λεπτό θα αρχίσουμε, γι' αυτό παρακαλώ καθίστε. Βολευτείτε και καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Should I wait slightly longer or not? Otwieram obrady. Συνεχίζουμε τις εργασίες της Ολομέλειας που διεκόπη στις 16 Ιουλίου του 2009. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στη Βέστερ Πλάτ στον εορτασμό της ε, ε, περτίου, ε, 20 από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θέρισε πολλά θύματα, εκατομμύρια θύματα στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει ουδέποτε να ξεχνούμε ότι η βία και ο πόλεμος μπορούν κάποια στιγμή να επανέλθουν στην Ευρώπη. Ε, γιατί τότε συνέβησαν και διάφορες άλλες ε, ε, βίαιες ενέργειες. Δύο ε, υπάλληλοι της πολιτοφυλακής της Ισπανίας δολοφονήθηκαν από την ΕΤΑ εν υπηρεσία. Με μεγάλη θλίψη επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για το θάνατο